Συνάδελφοι, παρακαλώ λίγη ησυχία για να συνεχίσουμε. Το άρθρο 191 του εσωτερικού κανονισμού προβλέπει για τις υποψηφιότητες με την επιφύλαξη του άρθρου 15 προβλέπει ψηφοφορία μυστική. Έγινε πρόταση από το Πρόεδριο να γίνει επί χάρτου η μυστική ψηφοφορία. Για ψηφοφορία με τις κάλπες. Όμως ο κανονισμός δεν το λέει αυτό Και η Ολομέλεια πάντοτε έχει το δικαίωμα να λάβει την τελική απόφαση. Γι' αυτό λάβαμε την, κάναμε αυτή την ψηφοφορία και θέσαμε σε ψηφοφορία ακριβώ τη διαδικασία με την οποία και θα προχωρήσουμε την ηλεκτρονική. Όλα αυτά με πλήρη σεβασμό τον όσο ορίζει το ο κανονισμό μα που το αναφέρει ρητό στο άρθρο 191, ότι η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τις εργασίες μα με τον τρίτο γύρο ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε, όπως είπα, ηλεκτρονικός. Καλώ όλους τους συναδέλφους να βάλουν την κάρτα ψηφοφορία τους στο μηχάνημα για να κάνουμε ένα τεστ, μια δοκιμή. Πρέπει να βεβαιωθούμε για το σύστημα. Καθώς είναι και η πρώτη ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου μετά από το διάλειμμα. Τεστ με πέντε τραγουδιστές. Θα δείτε τα ονόματα και με τον Γκένσορα μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. Επιλέξτε τον υποψήφιο με το γαλάζιο πλήκτρο κάτω δεξιά στην οθόνη. Παρακαλώ, ησυχία. Ή με τα πλήκτρα τα οποία μπορείτε να πατήσετε στα δεξιά. Ανάβει το γαλάζιο χωτάκι και βρίσκεται ένα αστεράκι δίπλα στα ονόματα. Και κάθε φορά που πατάτε ένα όνομα μειώνεται ο αριθμός των εδρών που πρέπει να κατανεμηθούν. Για να σεβαστούμε το μυστικό χαρακτήρα της ψηφοφορία. μετακινείται ο κένσορας, αλλά δεν φαίνεται πια ο αστερίσκος. Εάν είστε έτοιμοι, κάνουμε το τεστ με τους πέντε τραγουδιστές. Κυρίσουμε την έναρξη της ψηφοφορίας. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Vediamo i risultati. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Για να δούμε με τους τραγουδιστές τι έγινε. Είναι όλα ονόματα διασύμων. Το σύστημα λειτουργεί από ό,τι φαίνεται. Οπότε να περάσουμε στην πραγματική ψηφοφορία την οθόνη σα θα εμφανιστούν τα ονόματα των υποψηφίων. τρει. Μπορείτε να τοποθετήσετε τον κένσορα στο όνομα της προτίμησής σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Εψήφισαν άπαντες. Εψήφισαν άπαντες. περιμένουμε και εσάς, συνάδελφε. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εψήφισαν 411 βουλευτές. άκυρες ψήφοι 61, έγκυρες 350, εκλέγεται ο κύριος Καστάλντο με 248 ψήφους. Ο κύριος Κρασνοντεύσχη πήρε 85, η κυρία Μπιτζότο 17. Συγχαρητήρια στον κύριο Καστάλντο. Eh, Και τώρα για την εκλογή των κοσμητόρων του Ευρωκοινοβουλίου. Συνάδελφοι, προτείνω να ορίσουμε προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητων απόψε στις 22.10 το βράδυ. Οι υποψηφιότητε πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία στο ε, κτίριο Λουίς Βάη, στο γραφείο R00101 ε, και οι ψηφοφορίες θα γίνουν αύριο 4 Ιουλίου στις 9 το πρωί θα ξεκινήσουμε. Από τις 9 έως τις 11.30. Έχει δημοσιευτεί μερίσια διάταξη και στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου. Διακόπτεται η Ολομέλη. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας.